για δεύτερη ανάγνωση της εκθέσεως του κυρίου Λάιχτφριντ με έξαρση επιτρεπόμενες διστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην κοινότητα με την κυρία Τζουφρίντα πρώτα που ελπίζω να είναι εδώ Έχετε το λόγο κυρία Τζουφρίντα, ένα λεπτό Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπερψήφισα αυτή την σύσταση γιατί για την ασφάλεια όλων είναι σημαντικό τα βαρέα οχήματα και τα λεωφόρια που κυκλοφορούν εντός της Ένωσης να σέβονται συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά το βάρος, το ύψος, το μάκρος και το φάρδος τους. Και πάντοτε είναι θέμα ασφάλειας ε, το να παρέχονται και κάποιες εξαιρέσεις και να μπορούν οι παραγωγοί να κάνουν νέες προβλέψεις και προεκβολές ε, διότι η μηχανική μας επιτρέπει να βάζουμε καλύτερα οχήματα στους δρόμους μας ε, για να ελέγχεται καλύτερα ο αντίκτυπο σε περίπτωση σύγκρουση, καθώ και η τεχνολογία που μειώνει τι εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εμπορευμάτων που είναι ένα από τα σύμβολα της ΕΕ. Ευρώπης οπότε ας προστατεύσουμε την κατηγορία αυτή, ας βελτιώσουμε τις δύσκολες ε, συνθήκες εργασίας του και ας αυξήσουμε την ασφάλειά τους καθώς και τη δική μας κατά συνέπεια. Ευχαριστώ. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση και θα ήθελα να ζητήσω τους συναδέλφους που εγκαταλείπουν το ημικύκλιο κύκλιο, να το κάνουν σιωπηλά. Παρακαλώ ησυχία, παρακαλώ πολύ. Και δίνω το λόγο... Α, ο κύριος Κέλλη δεν είναι εδώ. Είναι? Α, συγγνώμη. Δεν είστε στη θέση σας, κύριε Κέλλη, γι' αυτό σας έχασα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Uh, Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά υπερψήφισα την ε, πρόταση αυτή συστάσεως, όπως και όλη η ομάδα μου. Είμασταν υπέρ των προτάσεων, πολύ σημαντικών προτάσεων και μάλιστα έγινε σήμερα το πρωί πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δρόμους ασφαλείς για όλους τους χρήστες. Και αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Επίσης, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούν να περιοριστούν οι κίνδυνοι αλλά και η επιβάρυνση των δρόμων μας από την υπερβολική ε, κυκλοφορία και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον προξενεί αυτή. Πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα βαρέα οχήματα, τα μεγάλα φορτηγά που χρησιμοποιούν τους δρόμους μας και πιστεύω με το κείμενο αυτό έχουμε την κατάλληλη βάση για να συνεχίσουμε τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση του κυρίου Λαμασούρ. Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά. Κεφάλαιο η κυρία Τζουφρίδα και πάλι. Σε αυτή τη φάση πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, από την οποία όλο και περισσότερο δυσκολευόμαστε να βγούμε, μία ε, είναι η βασική προτεραιότητα. Να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και οι μακροπρόθεσμε επενδύσει μπορεί να βοηθήσουν στην επιτύξη αυτού του στόχου, ε, χρηματοδοτώντα δραστηριότητε υλικέ όπω η κατασκευή υποδομών, όσο και αήλων όπω η ανάπτυξη έρευνα και τη ανάπτυξη, που είναι πολύ σημαντικέ για μακροπρόθεσμα γιατί αποτελούν ένα στοιχείο κλειδί για την ευφυή ανάπτυξη ώστε να αποφευθούν νέε κρίσει. Και η δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για μακροπρόθεσμε επενδύσει μπορεί να οδηγήσει στην μία μόνιμη ροή χρημάτων για όλου όσου ε, θέλουν να έχουν προτεραι... Ε, προοπτική μακροπρόθεσμα και σκέφτομαι του Δήμου και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Εάν επιθυμούμε να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το δημοσιονομικό στοιχείο, γιατί η Ένωση θα πρέπει να υποδείξει σε όλα τα μέλη ώστε να εισάγουν ε, φοροαπαλλαγή απαλλαγέ, ειδικά όσο, για όσου θέλουν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μάλαβιτ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Οι ε, μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές ε, είναι πολύ σημαντικές για την Ευρώπη, όπως και οι επενδύσεις. Ε, στην πρώτη γραμμή θα είναι ιδιωτικές επενδύσεις που επιτρέπουν την έρευνα και την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη προσπαθεί με διάφορους τρόπους να στηρίξει τις επενδύσεις και να αυξήσει το επίπεδό τους στα διάφορα έργα. Τα προγράμματα της Ένωσης, περνώντα από τα διαρθρωτικά ταμεία μέχρι τα νέα μακροπρόθεσμα, μάλλον ταμεία για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, έχουμε ένα ολόκληρο φάσμα απαραίτητων μηχανισμών για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Έτσι θα μπορέσουμε να διοχετεύσουμε νέες, ε, μάλλον να δρομολογήσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις προς όφελος του τομέα της ενέργειας των, των μεταφορών και θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε περισσότερες χρηματοδοτήσεις. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Καταψήφισα την έκθεση διότι η συγκεκριμένη έκθεση συντηρεί τις δομές και τις διαδικασίες οι οποίες έχουν οδηγήσει στην οικονομία καζίνο. Έτσι παρότι δόθηκαν 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωση των τραπεζών εντούτοις έχουμε είκοσι εκατομμύρια ανέργους στην ευρωπαϊκή ένωση γιατί τα κεφάλαια αυτά δεν δόθηκαν από τις τράπεζες για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας. ταυτόχρονα ενώ δόθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στις χώρες του μνημονίου τελικά το χρέος αυξήθηκε και μαζί και η ανεργία. στην ελλάδα παρότι δόθηκαν 214 δις ευρώ ως δάνεια τελικά έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην ανθρωπιστική κρίση και εκατομμύρια ανέργους. για να έχουμε λοιπόν επενδύσεις στην πραγματική οικονομία πρέπει με νόμο να επεκταθεί ο διαχωρισμός εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών να έχουμε μια νέα glass steagall act. ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Με χαρά υποστήριξα και αυτή την έκθεση. Για την οποία έγινε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση το πρωί. Ο εισηγητής κύριος Λαμασούρ έκανε καταπληκτική δουλειά. Πρέπει βεβαίω για να ξεφύγουμε από την ύφεση να γίνουν επενδύσει και κυρίω εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Ιδιαίτερα έχω υπόψη μου την ανάγκη σε σε βασικές ε, υποδομές μεταφορών και ενέργειας. Όπως είπα και νωρίτερα. Όπως αναφέρθηκε άλλωστε το πρωί, έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται και πάλι οι τραπεζές μας το 70% των ε, ιδιωτών που προσφέρουν σε αυτές για να εξασφαλίσουν δάνειο, το εξασφαλίζουν κιόλας. Και εάν συνεχίσουμε με αυτές τις επενδύσεις μπορούμε να ξεφύγουμε ασφαλώς από την ύφεση. Ευχαριστώ Πόλτσακ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ε, ευχηθώ στην Επιτροπή κάθε επιτυχία στην εκτέλεση των μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί η Ευρώπη χρειάζεται νέα ανταγωνιστική ανάπτυξη και καινοτομία. Χρειάζεται επίσης να θέσει σε εφαρμογή την πολιτική συνοχή της. Η οικονομία είναι κυκλική. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Εκφύσεως. Και άρα μετά την ανάπτυξη έρχεται περίοδος ύφεσης. Λογικός πώς. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μελλοντικές ε, με μεθοδολογικούς κλειδονισμούς έχοντας υπόψη τους κλειδονισμούς του παρελθόντος. Γι' αυτό και υποστηρίζω τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Γιατί βεβαίως μπορεί να βλέπουμε μόνο πώς ε, επέδρασαν οι κλειδονισμοί στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναδρομή στα δύο-τρία χρόνια περίπου. Θα πρέπει, η πρόεδρος διακόπτη, ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρώ στις ε, επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση του κυρίου Ταραμπέλα. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την έκθεση του κυρίου Ταραμπέλα για την ισότητα μεταξύ αδρών και γυναικών και θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί. Νομίζω ότι χάσαμε μια ευκαιρία να στείλουμε δηλαδή ένα σαφές μήνυμα σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη βελτίωση θέση των γυναικών, τη μεγαλύτερη εκπροσώπησή της σε πολιτικούς φορείς κτλ. Δυστυχώς το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέχει διατάξεις ή συστάσεις υπέρ των αμβλώσεων για παράδειγμα. Που θα είναι και μία μέθοδος αντισύλληψης όπως ε, τελικά φαίνεται να προωθείται. Αυτό για μένα είναι μια παραβίαση των δικαιωμάτων του αγέντου παιδιού. Επίσης, παραβιάζονται κανένα επικορικότητας από το Κοινοβούλιο, διότι αυτά είναι ζητήματα που τα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη ατομικά. Πώ πει ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ τάχθηκα υπέρ τη εκθέσεως για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και εάν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι στην πρώτο καθεδρία, στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οπωσδήποτε πρέπει να ταχθεί στο θέμα αυτό. Στο άρθρο 45 έγινε η συζήτηση ιδιαίτερα στο δικαίωμα δηλαδή των γυναικών να επιλέγουν, να κάνουν τι επιλογές ω προς την γενετήσια υγεία και κυρίως το δικαίωμα στην άμβλωση τη διακοπή της εγκυμοσύνης. Εγώ υποστήριξα αρχικά ένα άρθρο του ECR που θεωρούσε ότι θα πρέπει αυτό να υπαχθεί στην αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις στα θέματα αυτά. Άρθρο το οποίο δεν πέρασε. Αλλά υπερψήφισα τη διατήρηση του άρθρου 45 στο σύνολο του κειμένου. Γιατί θεωρώ ότι το δικαίωμα της γυναίκας στην αναπαραγωγική υγεία έχει πολύ μεγάλη σημασία όσο μεγάλη σημασία έχει και η χρήση των αντισυλληπτικών. Βέβαια είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και θα πρέπει σε επίπεδο κρατών μελών να επιλύονται. Κυρία Τζούφριντα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ταραμπέλα, την έκθεση το οποίο υπερψήφισα βεβαίω. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί την πλούσια έκθεση ε, αναφέρονται οι φραγμοί που πρέπει να ιτηθούν ώστε να αρθούν ώστε να αυξηθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μιλά για ανισότητα στου μισθού, στι συντάξει, στην απασχόληση, στην υγεία. Κανένα δεν ζητά υπηρεσίες για τι γυναίκε, Λείπει ένα σύστημα πρόνοια για όλε εκείνες τις κατηγορίες που φροντίζουν οι γυναίκε ω μητέρε, ε, αδερφέ. Ε, ε, λείπουν λοιπόν, οι κατηγορίε στι οποίε φροντίζουν οι γυναίκε, όπω οι ηλικιωμένοι. Θα πρέπει να θυμηθούμε λοιπόν να επενδύσουμε στην πρόνοια, στην αποτελεσματική πρόνοια την οποία αναλαμβάνει το κράτος για όλους, όχι μόνο για τις γυναίκες. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο την ευελιξία και την ανάπτυξη, γιατί πριν και πέρα από αυτά έρχονται οι άνθρωποι και τα δικαιώματά τους. Και καταρχήν αυτά των γυναικών για να μπορούν να ασκούν το επαγγελμά του χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν κάποιον και έτσι ώστε η κοινωνία να είναι στο ύψο τη γυναίκα. Δεν βλέπω την κυρία Μελίνα, άρα κύριος Λούκε. Καταψήφισα την έκθεση αυτή. Διότι πιστώ, πιστεύω ότι είναι ε, ύπουλο το να αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην άμβλωση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Όχι, το δικαίωμα, το ανθρώπινο είναι δικαίωμα στη ζωή και δικαίωμα στο απαραβίαστο του σώματος. Αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό από το να μπορεί η γυναίκα να αποφασίζει την άμβλωση, γιατί αυτό είναι μια ε, καταποκοπήν επιλογή που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι ντροπή να μπαίνει μέσα στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου φαίνεται αποτροπαίο το να γίνεται μια προσπάθεια με επικάλυψη τον τίτλο «Ανθρώπινα δικαιώματα» να περνάει μια παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εξού και καταψήφισα την πρόταση. Κυρία Μόρβα, έχει το λόγο ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ στην Ουγγαρία, την πατρίδα μου. Έχουμε πολλές γυναίκες εξατλημένες, σωματικά και ψυχικά κατεστραμμένες, με τις οποίες συχνά συνομιλώ. Είναι γυναίκες οι οποίες έχουν αναλάβει την ε, ανατροφή των παιδιών τους, ε, τη φροντίδα για τους ηλικιωμένους συγγενείς, και που επιπλέον καλούνται να δουλέψουν έξω από το σπίτι για να αποδείξουν ότι είναι γυναίκες αλλά ταυτόχρονα και εργαζόμενες πλήρους απασχόλησης. Πολλές φορές αναλαμβάνουν θέσει εργασίες που πληρώνουν πολύ λιγότερα από ό,τι τους άντρες συναδέλφου του. Εγώ υπερψήφισα το έγγραφο, διότι πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση αυτή τη τραγική κατάσταση. Αλλά το σύνολο δεν μπόρεσα να το εγκρίνω διότι αναφέρεται σε δικαίωμα στην άμβλωση αλλά κανένα μέτρο δεν προτείνει για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων. Η κυρία Τζεντήλ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εκτίμησα και συμμερίζομαι άρα το πολιτικό πλαίσιο αυτού της έκθεσης του κ. Ταραμπέλα. Ε, ωστόσο, θα πρέπει να μην μείνουμε σε μια ιδεολογική προσέγγιση, γιατί ο βαθμός του πολιτισμού ε, μετράται με την ε, ε, με βάση τα δικαιώματα αλλά και με την πρόνοια που προβλέπεται για τα πιο ευάλωτα άτομα που τη συναποτελούν, άρα και για τις γυναίκες. Ε, θα πρέπει να μπορέσουμε μέσω της πολιτικής μας να ξεπεράσουμε κάθε φοντομεταλλισμό όσον αφορά την ε, λαϊκή οπτική για αυτά τα θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να επιστηρίξουμε τα απελευθέρωση της ζωής των γυναικών, να αναγνωρίσουμε πως έχουν το δικαίωμα να ζήσουν τη σεξουαλικότητά τους χωρίς προκαταλήψεις, ακόμα και όταν είναι ενώπιον της της επιλογής να εγκαταλείψουν την εργασία τους ενώπιον μιας, ε, μιας μητρότητας ή ε, όταν πρέπει να εγκαταλείψουν ή μάλλον όταν τους, γίνεται, ε, τους αρνούνται μία μητρότητα. Θα, ευχαριστώ διακόπτη η Πρόεδρος. Θα πρέπει να γεννάμε θα ευχαριστω διακοπτε η προεδρος θα πρεπει να γενναμε πλουτο και όχι φτώχεια. Ευχαριστώ ο κύριος Σεντερχόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπόρεσα να υποστηρίξω την έκθεση αυτή. Αν και υποτίθεται ότι θα σημείωνε κάπου, κάποιο τρόπο κάποια τομή. Όμως αυτού του είδους η τομή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας και υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να παραμείνουν από τον έλεγχο των κράτων μελών. Για παράδειγμα, η αναπαραγωγική η σεξουαλική υγεία των γυναικών Έχω πει και θα το ξαναπώ. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η νομοθεσία της έχουν όρια, έχουν τα όρια τους. Δεν θα πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Merci. La parole est à Monsieur Morgano. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μοργκάνο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ε, πήγα στην, ε, στο ψηφι, στην ε, ψηφοφορία για το ψήφισμα του κυρίου Ταραμπέλ όσον αφορά την ισότητα ανδρών γυναικών για το 2013. Αν και πολλά πράγματα συμμερίζομαι, υπάρχει κάτι που, θέλει να επιβάλλει το δικαίωμα της αμβλωσής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετέτρεψε τη χθεσινή και σημερινή συζήτηση στην ουσία ως μια, έναν απολογισμό για την τραγωδία που μπορεί να είναι είναι μια δυνητική ε, ε, άδεια για την μάλλον απελευθέρωση της άμβλωσης ενώ θα έπρεπε να είναι μια συζήτηση για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των ε, γυναικών. Εάν δεν υπήρχε αυτό το επιπλέον στοιχείο θα μιλούσαμε για τα θετικά στοιχεία της έκθεσης αυτής που δεν λείπουν και επαναλαμβάνω ότι γι' αυτό και απήχα από την ψηφοφορία για το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Φορέντζα έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πως η σημερινή ήταν μια σημαντική ψηφοφορία που σαφώς ε, ήταν ευνοϊκή για το ψήφισμα Ταραμπέλα και εν μέρη βελτιώνει την άσχημη θέση που είχε, είχε κρατήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την απόρριψη δηλαδή της έκθεσης Εστρέλα. Πιστεύω πως σήμερα έχουμε βάλει στο επίκεντρο της συζήτησης ε, και στη συζήτηση της Ευρώπης την αυτοδιάθεση, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης κάθε γυναίκας και την ελευθερία των γυναικών και πιστεύω πως το κείμενο του Ταραμπέλα συμβάλλει στο να καταλάβουμε και να καταστήσουμε σε προφανές πως η δική μου γενιά ε, των γυναικών το γνωρίζει, πως η λιτότητα είναι μια, βασι... είναι μια η επίθεση στο δικό μας δικαίωμα δικαίωμα αυτοδιάθεση. Δεν θέλουμε εμεί νόμου για το σώμα τη γυναίκα, αλλά ένα σύστημα πρόνοια και δικαιωμάτων που θα μα αφήνει να επιλέξουμε και να έχουμε την αυτο... δικαίωμα αυτοδιάθεση. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για την ε, ε, πρόσκαιρη εργασία των γυναικών. Θα ήταν σκόπιμο να μιλήσουμε για ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κατά τη βία ε, που οφείλεται στο φύλλο. Θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα εμείς να αποφασίσουμε για το σώμα μας. Ευχαριστώ κύριο Σόγκορ. Ένα λεπτό. Διεθνή ημέρα για τη γυναίκα. Εάν θέλουμε να, επιβάλλουμε, να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων, όμω δεν αρκεί μόνο αυτό. Ένα βασικό ε, στόχο είναι η κατάργηση τη εμπορία των ε, ανθρωπίνων όντων που ε, κινείται από διάφορα κράτη-μέλη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το να είναι οι γυναίκε πιο οικονομικά ανεξάρτητε θα είναι λιγότερο εύκολο στόχο για την εμπορία. Ωστόσο, θα πρέπει να, αλλάξουμε, να λάβουμε υπόψη υπόψη και διαρθρωτικές λύσεις. Κάτι ακόμα που θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό ε, και συνδέεται με αυτή την έκθεση, συνδέεται με την ε, εκπαίδευση και την ε, παιδεία των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελόνης είχε προβλέψει κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα τα, σχετικά μέτρα είναι ανεπαρκή σε πολλές χώρες και στη δική μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Διότι φοβούμαι ότι εξωτερικοί εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν ε, την εσωτερική ιδιωτική ζωή των ατρών και των γυναικών. Και έχω και πολιτική μου ομάδα θεωρεί ότι οι οικογενειακές σχέσεις πρέπει να είναι συμβατικές παραδοσιακές. Δεν πρέπει να αλλάξουν στη χώρα μου, τη Βουλγαρία. Η οικογένεια είναι μια οικογένεια με έναν άντρα και με μια γυναίκα. Είμαι κατά οποιασδήποτε εξωτερική παρέμβαση από την Κομισιόν ή από άλλου θεσμού ε, και όργανα που εξώθεν θα επηρεάζουν τι οικογενειακέ ε, θέσει. Κάθε άνθρωπο έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσει που αφορούν την οικογένειά του και την υγεία του. Τα οικογενειακά προβλήματα και τα προβλήματα ανδρών και μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να τηρούν τις παραδόσεις, τις παραδόσεις πολλών αιώνων. Κύριο Σκέλη. Κυρία Πρόεδρε, με υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και μακάρι πάρα πολύ γρήγορα να ισχύει αυτό. Ταυτόχρονα είναι κρίμα στην ε, στο ψήφισμα αυτό να υπάρχουν συστάσεις, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, που έχουν να κάνουν ε, με την ε, καθιέρωση της άμπλωσης σε όλη την Ευρώπη. Είμαι κατά του ψηφίσματος, είμαι κατά αυτής της έννοιας της άμβλωσης που να επιτρέπεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσει κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Και στην προκειμένη περίπτωση γυναίκες γιατί αυτές αφορά οι άμβλες και όχι τους άντρες. Όταν όμως το θέμα αυτό το συζητήσαμε και όταν το ξανασυζητήσουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο πραγματικό θέμα της ισότητας. Και αυτό πρέπει να γίνει πολύ σύντομα. Πετήρ. Ευχαριστώ. Είμαι υπέρ της ισότητας μεταξύ όλων και μεταξύ των ίσων ευκαιριών για όλους. Δεν όμως, ε, δεν ε, προωθεί αυτής της αρχής η έκθεση. Ναι, μεν έχει ε, στον τίτλο του τη λέξη ισότητα, αλλά δεν εξασφαλίζεται ισότητα με το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Ξέρουμε ότι τέτοιου είδους εκθέσεις έρχονται σε αντίφαση με, και αντίθεση με αρχές βασικές όπως η αρχή της επικουρικότητας. Άρα, αν τη στηρίξουμε αυτήν την έκθεση, υπονομεύουμε τα θεμέλια και τι συνθήκε τη Ένωση και οδηγούμαστε σε ανασφάλεια δικαίου. Υπονομεύουμε το κράτο δικαίου. Δεν γίνεται ε, τελικά κατανοητό ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Ε, βλέπουμε αυξάνονται ανισότητε. Εγώ πραγματικά λυπούμαι, θλίβομαι που βλέπω ότι μια έκθεση που αποτίθεται ότι προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών γίνεται μια έκθεση η οποία κάνει διαφήμιση της άμβλωσης. Είναι, ε, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά της Ευρώπης. Ε, περνάμε τώρα στι επεξηγήσεις ψήφου της έκθεσης για τον ανταγωνισμό μέσα Σμιτέ. Ho votato a favore perché la η κυρία Τζουφρίδα, εγώ υπερψήφισα γιατί η ανταγωνιστικότητα είναι μια από τι συνταγέ για να βγούμε από την κρίση. Μια επαρκή αποτελεσματική ανταγωνιστική πολιτική θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα και την ευημερία των συμπολιτών μα. Ε, ενιαία αγορά για την, ενέργεια, για την ενέργεια, για τον οικονομικό τομέα, για την βιομηχανία, για τι μεταφορέ. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε και να προσέξουμε τη μεγάλη ευκαιρία που μα προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά χωρί να ξεχνάμε όλα τα σχετικά θέματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν πρέπει να είναι η μόνη αρχή που θα διέπει την δημιουργία και την εξέλιξη των αγορών. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή όταν υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο ο συντονισμό των πρωτοβουλειών, γιατί στον, την ανταγωνισμό θα πρέπει να τον συνοδεύει η απασχόληση και η ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπόρζαν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 Ο ανταγωνισμός ε, παρουσιάζεται ως ένας βασικός παράγοντας ανάπτυξης ε, για την Ευρώπη. Πάνω από το 20% ωστόσο των καταναλωτών διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να αγοράσουν online ε, πέρα από τα σύνορα. Το ηλεκτρονικό συνοριακό εμπόριο δεν αποτυπροσωπεύει παρά το 4% του εμπορίου. Αν θέλω να αγοράσω παπούτσια από την Εστονία, ο σερβερ μου λέει πως αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Όχι εσείς. Εάν αγοράσω ένα κάτι μια ηλεκτρονική συνδρομή ας πούμε και μπω σε μια γειτονική χώρα με μπλοκάρει για την πρόσβαση σε αυτό που ωστόσο έχω, έχω πληρώσει. Αυτά είναι καθημερινά παράπονα των συμπολιτών μας ενώ υπάρχουν περιπολικά αιτήματα ε, για τα οποία δεν μπορούν να απαντήσουν οι ε, εκτός ένωσης ε, έμποροι. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε μέχρι ότου να έχουμε ενιαία αγορά χωρίς διακρίσεις. Ο κύριος Μαριάς ο ανταγωνισμός υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη σημερινή φάση της λιτότητας και της φτώχειας στην ευρώπη. όμως για να λειτουργήσει ορθά ο ανταγωνισμός θα πρέπει να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ που υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα. επίσης πρέπει να καταδικαστούν πρακτικές φορολογικού ντάμπινγκ όπως η πολιτική juncker με τα γνωστά luxleaks ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να επιδείξει προσοχή στις συγχωνεύσεις προκειμένου να μην δημιουργούνται ολιγοπωλιακές συνθήκες και αυξάνονται οι τιμές. πρέπει τέλος να υπάρξει σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας χτύπημα του αθέμητου ανταγωνισμού και αύξηση των αρμοδιοτήτων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. καθώς οι σκέψεις αυτές ενυπάρχουν στην έκθεση την υπερψήφισα. ευχαριστώ. Ε, για ένα λεπτό. ευχαριστώ. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός των αγορών είναι μία από τις δυνάμεις ε, της κινητήριας για την δημιουργία και την καινοτομία. Αλλά υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, επιλογές και πρακτικές που ακολουθούν τα κράτη-μέλη, κατακαιρματίζοντας έτσι την ενιαία αγορά. Και δημιουργώντας προβλήματα και στον ανταγωνισμό, δημιουργώντας μονοπόλια τα οποία, στα οποία αντιστοιχεί το 3% περίπου του ΑΕΠ της Ένωσης. Η ε, πολιτική του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρωτώ αν επαρκεί για να υποστηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές φορές τις τιμές τις ορίζουν διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών με επιδοτήσεις ή ε, φορολογική, φορολογικά κίνητρα. Πρέπει λοιπόν αυτά να τα δούμε σαν ενθάρρυνση και όχι, πρόσβαση, και όχι δυσκολίες πρόσβαση στην αγορά. Η κυρία έτσι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υποστήριξα την ε, έκθεση του συναδέλφου Μέσσερ με την ε, επιλογή της ε, καλύτερης πρόσβασης στην αγορά ως προϋπόθεσης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το γεγονός ότι κάποια κράτη παρουσιάζουν απελευθέρωση μόνο επί χάρτου και διατηρούν ακόμη και μάλιστα με κυρίαρχη, με δεσπόουσα αγορές, ε, δημόσιες επιχειρήσεις ε, σε όρους μονοπωλίου που καταστρέφουν τις ε, συνθήκες του ανταγωνισμού και άρα μας οδηγούν σε μια παράλογη κατάσταση. Ο φορολογούμενος ωφελείται κατά τα φαινόμενα από μια υπηρεσία σε χαμηλότερη τιμή, αλλά με την υποχρεωτική συνδρομή του οδηγεί σε απώλειες. Οδηγείται τελικά σε απώλειες οικονομικές ενία αγορά πρέπει να εξασφαλίσει κανόνες ισότιμους για όλους. Ευχαριστώ κύριο Σιόνι, έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ως σοσιαλδημοκράτης ε, βουλευτής και σκιώδης εισηγητής υπερψήφισα την έκθεση θεωρώντας ότι μπορούμε να προσφέρουμε μια ακόμη ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου προστασίας των θέσεων εργασία και εξασφάλισης ε, καλύτερων υπηρεσιών. Ωστόσο ούτε εγώ ούτε η ομάδα μου μπορούμε να δεχθούμε τις προτάσεις για την ιδιωτικοποίηση στον χώρο των μεταφορών επί παραδείγματι που λέει η Άλτερ. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε το σημείο 85 της εκθέσεως. Γι' αυτό τελικά δεν δεχόμαστε με το σημείο αυτό, αλλά στο σύνολο υποστηρίζουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε σε επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Σάλμπα Μπιντεγκάιν, ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το λόγο έχει η κυρία Λόπε Μπερμέχου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταψήφισα την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί δεν θεωρώ ότι οι δράσεις της ε, ε, αξίζουν να τις δώσουν νομιμοποίηση και να την υποστηρίξει το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στήριζει κανονικά η έκτητα τα κράτη για να ε, περάσουμε μέτρα ανάκαψη οικονομίας, ε, θα πρέπει να φέρει σταθερότητα στις καταθέσεις, να στηρίξει ε, τα ομόλογα δημοσίου. Όμως τελικά με το ένα χέρι ο Ντράγκη <clears throat> τροφοδοτεί τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών φουσκών, ενώ κλείνει τη στρόφιγγα πίστη στα, που, στα κράτη που αγωνίζονται για τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι πιο διακριτική η μέθοδος από ότι η μέθοδος Τρισέ που ζητούσε περικοπές ή εργασιακές μεταρρυθμίσεις, αλλά με τις σημερινές μας ψήφους δείχνουμε για μια ακόμη φορά ε, τα μεγάλα κόμματα δείχνουν ότι προτιμούν ε, τα οικονομικά και συμφέροντα παρά την αλληλεγγύη με τον Ευρωπαϊκό Λαό. Κυρία Τσουφρίντα, για ένα λεπτό. Αυτή η έκθεση τονίζει και φωτίζει τις πτυχές που χαρακτηρίζουν τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα τελευταία χρόνια. Εκτιμούμε τις μη συμβατικές ε, ε, πολιτικές ε, που χρησιμοποίησε. Πέρα από τη σταθερότητα του τιμών, μέσα στις προτεραιότητες της έκθεσης θα πρέπει να είναι στόχοι όπως η ανάπτυξη και η επασχόληση. Βέβαια όλα αυτά δεν αρκούν σε σχέση με τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Θα πρέπει να παράλληλα να προχωρούν διορθωτικές μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις. Νομίζω πως είναι θετικό σημαντικό στοιχείο και η δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τη στιγμή που με δυσπιστία, αν όχι και με εχθρότητα βλέπουν οι πολίτες τα θεσμικά όργανα ήταν απαραίτητη μια προσπάθεια διαφάνειας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την κυρία Πάγκα Ο κύριος Μαριάς. Καταψήφισα την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2013 διότι η έκθεση αποδέχεται και επικροτεί το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα έχει μετατραπεί πλέον σε κράτος εν κράτη και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην περίπτωση της ελλάδας καθώς ο ντράγκη κατά παράβαση της συνθήκης ασκεί εκβιαστική πολιτική απέναντι στον ελληνικό λαό. ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπερψήφισαν μαζικά την τροπολογία που υπέβαλα. με την υπερψήφιση της τροπολογίας αυτής το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ζητά να σταματήσει η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει στο πλαίσιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας καθώς θεωρεί πλέον ότι η ect δεν μπορεί να είναι μέλος της τρόικας και ταυτόχρονα να ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη νομισματική αρχή. και αυτή η εξέλιξη είναι ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να πετάξουμε την τρόικα έξω από την πατρίδα μας στην ελλάδα δικαιώνοντας έτσι την ψήφο του ελληνικού λαού στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η πιστωτική ασφιξία που επιβάλλει ο ντράγκη στην ελλάδα δεν πρόκειται να περάσει. ο αγώνας συνεχίζεται. Uh, εγώ υπερψήφισα όλες αυτές τις ε, προτάσεις και όφιλα να το πράξω γιατί βρίσκομαι εδώ Μάλλον, γιατί ακούω ότι ο πρόεδρος Ντράγκη παρουσιάζει αυτή την πρόταση και πιστεύω πως η δική μας ψηφοφορία εδώ ε, θα ε, ενισχύσει τα όσα με αυτή τη συζήτηση και πρέπει λοιπόν να επενέσω την εργασία του. Καλωσορίζω όλα όσα υπόθηκαν στην έκθεση, αλλά θα πρέπει επίσης να πω ότι υπάρχει ένα άλογο, κούρσες, ε, που ε, λέγεται ποσοτική χαλάρωση. Εγώ έχω ποντάρει σε αυτό το άλογο που τρέχει στον αγώνα. Ελπίζω πως θα έρθει πρώτο και ότι θα είναι ε, τόσο επιτυχές όσο και ο κύριος Ντράγκη μέχρι ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Μακάρι να κερδίσει πολλά ε, εκεί που έχει ποντάρει ο κύριος Κέλλη. Αλλά η της έκθεση της του 2013 είναι το θέμα μας και θα ήθελα να στηρίξω με την ευκαιρία τα βήματα και τα μέτρα που λαμβάνει η έκτη. Έχει ξεκινήσει μια επικίνδυνη προσπάθεια ταξίδι να περιορίσει τους τεράστιους κινδύνους λόγω αποπληθωρισμού που θα μπορούσε στην Ευρώπη να οδηγήσει σε μια περιδίνηση. Και αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι οι αποπληθωριστικοί κίνδυνοι δικαιολογούν απόλυτα τα μέτρα αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό και αξίζει να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Νομικών Υποθέσεων.